Ιράν και θα ζητούσα από τη διάσκεψη των Προέδρων που έδωσε το πράσινο φως στην αποστολή αυτή ε, να αναθεωρήσει την απόφασή της διότι δεν θέλουμε να στηρίξουμε την κυβέρνηση του Ιράν. Ευχαριστώ. Ε, εγκρίνονται τα πρακτικά της 29ης Σεπτεμβρίου και εφόσον, εφόσον δεν υπάρχει κανένα σχόλιο περί αυτών. Λοιπόν, Κυρίες και κύριοι, έχω την ακόλουθη ε, ενημέρωση. Θέλω να καλωσορίσω μία αντιπροσωπεία από το Κοινοβούλιο του Λιβάνου επί τους κυρίους Καμπάνη, Μπάζη και Μπακραντούνιαν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στη σχέση με το Λίβανο διότι πολλά από τα κράτη-μέλη συμμετέχουν στην αποστολή ε, Φινούλ και ε, ε, το, ο Λίβανος είναι μία από τις σπάνιες αραβικές χώρες οι οποίες έχει δεχθεί ε, μία αποστολή εκλογικής παρατηρήσεως Ευρωπαϊκής Ενώσεως θέμα που απασχολεί πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις, για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο με αυτά κοινοβούλια και σας ε, καλώ να ε, προωθήσετε αυτές τις ε, τακτικές ανταλλαγές. Ελπίζω ότι οι συνεδριάσεις και οι συναντήσεις που είχατε χθε και σήμερα ήταν ε, επικοδομητικές και ότι η παραμονή σας στις Βρυξέλλες θα τίνει στη βελτίωση των ε, δύο θεσμικών οργάνων μας. Σας ευχαριστώ. Έχω να σας δώσω και δύο επιπλέον πληροφορίες. Καταρχήν, Έχουμε καλά νέα αλλά και ανησυχητικά νέα από τον νότο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θέλουμε να χαιρετήσουμε τη σταθεροποίηση της καταστάσεως στη Λιβύη αλλά μας ανησυχεί η ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων και η Τινησία ε, θα οργανώσει τις πρώτες ελεύθερες εκλογές της γι' αυτό και σε λίγες εβδομάδες θα επισκεφθώ τη Λιβύη και την Τινησία να εκφράσω τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία εκδημοκρατισμού και τη δημιουργία μιας ελεύθερης αγοράς καθώς επίσης και τη μελλοντική ε, συνεργασία ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τη Λιβύη και την Τινησία. Πρέπει να σταματεί η περιοχή αυτή και αντιθέτως οι στρατιωτικές αρχές θα έπρεπε να ενθαρρύνουν και να συγκρατήσουν ε, το λαό ε, ε, εγγυόμενοι την ελευθερία των θρησκευτικών μειονοτήτων διότι υπάρχουν ακόμη βία σε διάφορες από αυτές τις χώρες εναντίον του ιδίου του λαού τους και πρέπει να ενθαρρύνουμε την τους πολίτες ε, να καταστήλουν ε, ε, αυτή την καταπίεση και να εκδημοκρατιστούν. Επίσης με μεγάλη ανακούφιση με μεγάλη μάλλον λύπη ακούσαμε την τιμιγορία κατά της κυρίας Τιμοσέγκο πρώην Πρωθυπουργού της Ουκρανίας σε 7 χρόνια κάθυρξη και μας ανησυχεί η, ε, ε, η ε, διαφάνεια του δικαστικού σώματος και η ανεξαρτησία του διότι ετοιμαζόμαστε στο τέλος του χρόνου να συνάψουμε μία συμφωνία συνδέσεως με τη χώρα αυτή και καλούμε την ε, κυβέρνηση να ε, σεβαστούν τις αρχές οι οποίες διέπουν το πνεύμα της συνεργασίας μας. Κυρίες και κύριοι, έχω να κάνω και άλλες ανακοινώσεις η κυρία Λένα Εκ μου είπε ότι ε, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 και 4 ε, έχει ε, κληθεί να συμμετάσχει στην κυβέρνηση της Σουηδίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει ότι έχει κενωθεί η θέση της από τις 29 Σεπτεμβρίου. Επίσης όσον αφορά ε, την ε, δήλωση, γραπτή δήλωση 27 του 2001 στην αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Παλαιστινιακού κράτους η οποία ε, δεν έχει πλέον αντικείμενο εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε το ψήφισμα της 29 Σεπτεμβρίου 2011 για την κατάσταση στην Παλαιστίνη και απεσήρθη από τους συντάκτες της και τώρα επανέρχομαι η στην ημερήσια διάταξη η οποία υιοθετήθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων στις 29 ε, Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τον ε, εσωτερικό κανονισμό και ε, οι ε, επόμενες αλλαγές έχουν συμφωνηθεί. Ε, σήμερα, ε, Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, καταρχήν όσον αφορά τη συζήτηση για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23 Οκτωβρίου, τα ψηφίσματα θα υποβληθούν, σχέδια ψηφισμάτων θα υποβληθούν και οι προθεσμίες είναι ως εξής για προτάσεις ψηφισμάτων 12 το μεσημέρι 3η 11 Οκτωβρίου τροπολογίες και κοινέ προτάσεις ψηφισμα... ψηφίσματος 10 το πρωί Τετάρτης 12 Οκτωβρίου οι τροπολογίες της προτάσει ψηφισμάτων 11 το πρωί 12 Οκτωβρίου όλες αυτές οι προθεσμίες έχουν λήξει και όσον αφορά τις χωριστές ψηφοφορίες, έχετε χρόνο σήμερα μέχρι τις 7 το απόγευμα ε, για να υποβάλλετε τις προτάσεις σας και αυτό έχει συμφωνηθεί με όλες τις πολιτικές ομάδες. Η συζήτηση για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και Ρουμανίας στον χώρο του Σέγγεν θα περιλάβει και ε, προφορικές ερωτήσεις από τους φιλελεύθερους την Ηνωμένη Αριστερά και ε, τους Ευρωπαίους Ομοσπονδιακούς Δημοκράτες. Η,